Συγγνώμη, πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρτη, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37. άρχιτη ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 38. άρχιτη ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εκτιμώντα Ι. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Έκθεση Φωτίγα. Τροπολογία 1. Άρχεται η σοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1Q. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1S. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για κυρία Φώτιγα. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, μα έγινε ένα προφανές τεχνικό λάθος. Αναφερόμεθα στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Και γι' αυτό προτείνω να απαλείψουμε τις λέξεις ε, επόμενη, next και η διάδοχός της. Γιατί τώρα ε, αναφερόμεθα στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ, έχει κανείς κάνει αντίρρηση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 1AG. Αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση. Δεν σήκωσαν όλοι το χέρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Ψήφισμα ε, σύσταση στο σύνολό της, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Έκθεση Λόπες Αγγιλάρ. Τροπολογία 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. άρχιτε ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. άρχιτε ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. άρχιτε η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Διακόπτουμε για μερικά λεπτά και ξαναρχίζουμε αργότερα με τις επεξηγήσεις ψήφου.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 Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στι ιτολογήσει ψήφου. Έχω λάβει πολλά αιτήματα. Δεν μπορούμε όμως να πάμε πέρα από τις 14 και 45 προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεδρίαση η σύνοδος στις 3 το μεσημέρι. Επομένως, Όλες οι αιτιολογήσεις ψήφου είναι απομείνασες, θα εξεταστούν αύριο μετά την ψηφοφορία. Άλλες αιτιολογήσεις ψήφου θα μπορούσαν επίσης να υποβληθούν και γραπτός. Ας περάσουμε τώρα πρώτα στην σύσταση Φώτιγκα. Ο κύριος Πόσπισιλ έχει πρώτος το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα αυτήν την ε, εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση της χώρας και να βρει μια ε, διέξοδο από τον εμφύλιο πόλεμο. Ε, είμαι περήφανος που εκατοντάδες Τσέχοι από τη χώρα μου συμμετέχουν στην αποστολή ειρήνευσης στο Αφγανιστάν. διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτή την έκθεση και ελπίζω να είναι ένα βήμα στο δρόμο προς την ειρήνευση του Αφγανιστάν. Επιτέλους να υπάρξει κάποιος συμβασμός με τους Ταλιμπάν. Αλλά δεν ξέρω πόσο είναι πιθανό. Θα είναι πολύ δύσκολο παρόλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ τώρα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Και εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης να συναυθεί αυτή η συμφωνία γιατί νομίζω ότι όντως είναι σημαντικό να βοηθήσουμε την χώρα αυτή να αναπτυχθεί γιατί οι καταστροφές που έχει υποστεί ε, είναι κάτι το οποίο εμείς προκαλέσαμε και τώρα ε, ε θερίζουμε τους πικρούς καρπούς και οι επιπτώσεις ε, είναι και στις χώρες μας. Πρέπει να στηρίξουμε τους Αφγανούς που καταπολεμούν την ε, τρομοκρατία αλλά και την τρομερού επίπεδου εμπορία ναρκωτικών και δεν στηρίζουμε μόνο τους, ε, ε, τους στρατιώτες μας για να υπάρξει κάποιο είδους ειρήνευση αλλά για να υπάρξει κάποιο είδους πρόοδο στη χώρα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι όντως πρέπει να στηρίξουμε την ε, αφγανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εξυγχρονίσει τη χώρα για να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες. Γιατί μόνο με αυτά ε, ωφέλη θα πιστεί ο λαός του Αφγανιστάν να προχωρήσει στην ειρήνη. Ο κύριος Χάναν, και εσείς ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Αφγανιστάν ε, ανάλογα με όλες τις ταξινομήσεις των Ηνωμένων Εθνών είναι από τα πιο ε, διεφθαρμένα και φτωχά τμήμα, τμήματα της Ιφιλίου. Ε, γιατί όμως, δεν θέλω να υπεραπλουστεύσω, έπαιξαν ε, διάφοροι παράγοντες ρόλο, αλλά τουλάχιστον ένας ε, παράγοντας είναι ότι ποτέ δεν ήταν εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε ένα ένα έθνος που να αποτελεί τη δημογραφία της χώρας. Υπάρχουν Τατζίκοι, Ουσμπέκοι, Παστού και άλλοι. Δημιουργήθηκε τεχνητά ως ένα κράτος μαξιλαράκι. Και γι' αυτό η ιστορία είναι μια σειρά από πραξικοπήματα, δικτατορίες, επαναστάσεις και εισβολές. Ε, μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις ε, την ε, τελευταία 50 ετία είναι η δημιουργία πολλών νέων εθνικών κρατών. Από τα 180 έχουμε περάσει 230 κράτη-μέλη την τελευταία αυτή περίοδο και αυτό έχει οδηγήσει σε περισσότερη δημοκρατία και ευημερία πολύ δυστυχές ε, που διαπιστώνουμε ότι αυτή η χώρα πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αυτό όσον αφορά τη σύσταση, τώρα αιτιολογήσεις ψήφου για την έκθεση Φώτιγκα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λοιπόν, για την έκθεση έλεγα, Φώτιγκα, παρακαλώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινήσατε τις επεξηγήσει ψήφου με την έκθεση Φωτίγκα. Αλλά η έκθεση του κ. Στρογεύσκη για το πρόγραμμα έρασμο και το ε, σκληρό Brexit ε, προηγήθηκε. Δηλαδή θα καλύψω αυτό το θέμα, θα έχουμε επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Στρογεύσκη. Εγώ ζήτησα να μιλήσω για την έκθεση Στρογεύσκη και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι στη μέση διάταξη. Ε, Κοιτάξτε, όσον αφορά την έκθεση Στρογεύσκη, δεν προβλέπεται εδώ πέρα δήλωση, αιτιολόγηση ψήφου, γιατί δεν συζητήθηκε ποτέ η έκθεση αυτή, άρα δεν προβλέπεται και τα λόγηση ψήφου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την έκθεση Φωτίγκα, ο κύριο Μέσερμιτ, για ένα λεπτό πρώτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω τον λόγο για το Αφγανιστάν όχι γιατί θέλω να κάνω επιπλέον μια ζήτηση για το θέμα αυτό ε, ή γιατί θέλω να προκαλέσω μια νέα επέμβαση. Όχι, εγώ θέλω να ασχοληθώ με ένα βασικό θέμα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δημιουργηθεί ένας ε, ευρωπαϊκός στρατός και αυτό στηρίζεται και από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Φαίνεται ότι οι πολλοί θεωρούν ότι εμεί πρέπει να λάβουμε πολύ ευρύ αρμοδιότητε στον τομέα ε, άμυνα. Η έκθεση Φωτίγκα μιλάει περισσότερο για ε, την συμβολή του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ε, συνδέει τις ΗΠΑ με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αυτό θέλουμε να συνεχίσει να παίζει το ρόλο. Δεν θέλουμε νέα αμυντικά μοντέλα με βάση το δόγμα Juncker. Δεν θέλουμε να είμαστε εμεί ε, ένα ε, νέο φορέα στρατιωτικό. Όχι, αρκεί το ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην έκθεση Λό και Γκάρντα. Λούσι Άντρεσον, για ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Άντρεσον έχει το λόγο. παρόλο ότι κανεί δεν ε, διαφωνεί με την ανάγκη καλύτερων ε, ευρωπαϊκών νόμων για να σωθούν ζωέ. Αυτή η πρόταση είναι απογοητευτική. Η Βρετανική κυβέρνηση ε, κατάφερε να αποδυναμώσει το κείμενο και θα πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό. Αποκλείστηκαν, αποκλείστηκε η υποχρέωση ε, πρόσβαση, ελεύθερης πρόσβασης στα μέσα και στα κτίρια. Από την άλλη μεριά βελτιώνονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ε, παράδειγμα τραπεζικές υπηρεσίε και άλλα σημεία και ε, αυστηροποιούνται οι ποινές, καθώς επίσης και ε, βελτιώνεται η εκπροσώπηση των αναπήρων. Γι' αυτό ψήφισα υπέρ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπισιλ τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Βέβαια τώρα θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο αισιόδοξη σε κάποια τη σημεία, πάντως ακολουθεί τη σωστή άγουσα θεωρώ. Δηλαδή λέει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίε και θα πρέπει να παράσχει υπηρεσίε στο πλαίσιο τη ευρωπαϊκή αγορά και οι υπηρεσίε αυτέ θα πρέπει να είναι προσβάσιμε για τα άτομα αναπηρίε. Νομίζω ότι η αρχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να στείλουμε το σημαντικό αυτό χειρομήνυμα, γι' αυτό το λόγο υπερψήφισα την έκθεση αυτή, μολονότι, όπω σα είπα, θα ήταν καλύτερο να ήταν λίγο πιο φιλόδοξη σε κάποια τη σημεία και να προβλέπει καλύτερη προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Ελπίζω ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα επανέλθουν στην έκθεση αυτή, βελτιώνοντα του όρου και τι προποθέσει προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίε, για προϊόντα και υπηρεσίε που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ τη έκθεση αυτή. Για ποιο λόγο, επειδή πιστεύω πως ε, η προσβάσιμη Ευρώπη θα είναι προς όφελο όλων. Είναι ένα ιδανικό, ένα όρομα, δεν θα πρέπει να έχουμε εμπόδια στην ζωή των πολιτών μας και όπου υπάρχουν θα πρέπει να έρονται. Αυτή η έκθεση βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την αναλογικότητα. Το κατά πόσο δηλαδή ορισμένε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να τηρήσουν όλες τις ε, απαιτήσει του κειμένου αυτού. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ιστοσελίδε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει απαραίτητα να τηρούν όλες αυτές τις απαιτήσεις. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χάναν ήθελε το λόγο, αλλά δεν το βλέπω στην αίθουσα, άρα ας περάσουμε στην έκθεση Κουέλιο. Η κυρία Μακοβέη πρώτη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το σύστημα VIS, το σύστημα για τις πληροφορίες για τις θεωρήσεις μας βοηθάει να δώσουμε θεωρήσεις και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές για το άσυλο, τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων να εξακριβώνουν πολύ σύντομα ποιοι πολίτες τρίτων χωρών εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης. Το νέο σύστημα VIS βελτιώνει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί με ευφυή τρόπο και να γίνεται η πρόθεση των δεδομένων ε, ταχύτατα. Η προστασία των εξωτερικών συνόδων τη Ένωση και η διαχείριση τη μετανάστευση και η βελτίωση τη εσωτερική ασφάλεια είναι τρία ουσιώδη στοιχεία. Ουσιώδη για όλου. Ο νέο κανονισμό εισάγει υποχρεωτικό χαρακτήρα για την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών από 6 ετών. Έτσι μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητα ενός παιδιού που ζητάει μια προξενική θεώρηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να εξακριβώσουμε ποια παιδιά έχουν κλαπεί. Ευχαριστώ κύριος Μέσος με ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η προστασία της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και τα τελευταία χρόνια είδαμε τι καταστροφές είχαμε, τι προβλήματα δημιουργήθηκαν δεν ε, ανταποκρίνονται οι πολιτικές στα προβλήματα των πολιτών. Είχαμε τον πόλεμο στην Συρία, είδαμε πώς οι τρομοκράτες μπαίνουν στη χώρα μας ως συνέπεια. Βλέπουμε πώς τα ανοιχτά σύνορα στη, στο εσωτερικό της Ευρώπης επιτρέπουν στα άτομα αυτά να πάνε παντού στην Ευρώπη και να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες. Τώρα δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε το πρόβλημα και για να καταφέρουμε να το επιλύσουμε το σύστημα αυτό είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι φτάνει πολύ καθυστερημένα. Πού θα ήταν η Ευρώπη σήμερα, αν χώρες όπως η Δανία και άλλες δεν είχαν ε, επανέλθει στους ελέγχους στα σύνορα. Θα είχαμε ακόμη περισσότερα προβλήματα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση Ντάλι. Ο κύριος Μέσερμιτ έχει πρώτο το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Λοιπόν, για τους περισσότερους Ευρωπαίους θα πρέπει να είναι σαφές. Οι Ευρωπαίοι δεν επιθυμούν το Κοινοβούλιο, οι διάφοροι οργανισμοί της Ένωσης, η Επιτροπή να αποφασίζουν για τη σύνθεση του πληθυσμού των χωρών μας. Αναμφίβολα, αυτό είναι το πιο βασικό θέμα. Γιατί θα δείξει πώς θα εξελιχθούν οι χώρες μας σε μία ή δύο γενιές με τις νέες ε, νοτροπίες ε, που μπορούν ε, να, μπούμε, να μπουν στις χώρες μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε εργαστήρια για μίξη πληθυσμών. Δεν είναι λοιπόν αυτή η καλή πρόταση. Η μόνη καλή πρόταση είναι το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει μόνο του την πολιτική του για το θέμα της μετανάστευσης. Αν μια χώρα έχει μια πλειοψηφία τη αριστερά, μπορεί να κάνει αριστερή μεταναστευτική πολιτική. Αλλά δεν μπορείτε να μα το επιβάλλετε παντού. Δεν είναι αυτό που επιθυμούν οι Ευρωπαίοι. Η κυρία Σίλβια Κώστα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτό το νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης ε, με το προπολογισμό αυτό των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει πολλές νέες καινοτομίε. Υπάρχει νέα αρχή της αλληλεγγύης στη νομική βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έφανση όσον αφορά την ένταξη και την ενσωμάτωση. Πέρα από το πρώτο στάδιο τη υποδοχή, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την αλληλεγγύη και την οικονομική ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί στο επίπεδο αυτό ότι θα τηρήσουν οι υπόλοιπε κυβερνήσει και η Ιταλική κυβέρνηση όλου ιδιαίτερω τι δεσμεύσει του στι χρηματοδοτικέ. Γιατί βλέπουμε ότι η Ιταλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μειώνει τη χρηματοδότηση όσον αφορά την υποδοχή, όσον αφορά την ένταξη, όσον αφορά την αλληλεγγύη. Σα ευχαριστούμε. κύριο Τζαμπάσκι τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα κατά του κειμένου. Παρόλο ότι η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σοβαρά σημερινά προβλήματα, η πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Πάλι προσπα... μιλάμε για την ένταξη των μεταναστών αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Και μιλάμε για ένταξη και των νομίμων και των παράτυπων μεταναστών. Το να ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούμε την ένταξη ατόμων τα οποία έχουν μπει παράνομα στην επικράτειά μας είναι κάτι απαράδεκτο για μένα. οι, η, διαβου, η, μικρο, η μη κυβερνητικέ ε, ε, οργανώσει που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο μεταναστών ήταν αυτέ που πιο πολύ συμμετείχαν στη διαβούλευση. Για να διαχειριστούμε την μεταναστευτική κρίση πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας σε βάθος. Ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη πολιτική βούληση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες και ανθρώπινες ζωές και να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο. Η δημιουργία του Ταμείου Μετανάστευση αποτελεί ένα πρώτο βήμα για αυτή την ανεθεώρηση μεταναστευτική πολιτικής μας. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, τα κράτη-μέλη θα ενισχύσουν και θα αναπτύξουν όλες τις πτυχές του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ε, θα αναπτύξουν ε, κανάλια νόμιμης μετανάστευσης για των χωρών, θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική και, αποτελεσματικές και βιώσιμες επιστροφές επαναπατρισμού των μεταναστών με την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής του φορτίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεταναστευτική κρίση αποτέλεσε σεισμό για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Η πολιτική ασφάλεια στις διάφορες ε, χώρες ε, στριμώχτηκε και μερικές, ορισμένες χώρες θεώρησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τους επιβάλλει μια συγκεκριμένη πολιτική. Η Σλοβακία ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης με ένα σύστημα το οποίο δεν θα αποτελεί μαγνήτη πόλο έλξης για τους ε, μετανάστες. Οι προσφυγικοί καταβλισμοί αυτή τη στιγμή ε, ε μια επίσκεψη στους προσφυγικούς καταβλισμούς θα ε, σας δείξει ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μείνουν εκεί. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας θα πρέπει να ε, μην εμπλεκόμαστε στις εθνικές αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην έκθεση Φαγιών. Ο κύριο Τζαμπάσκη έχει το λόγο. Το λόγο, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, σας παρακαλώ, σας ακούω. Μα και εγώ ζήτησα να κάνω επεξήγηση ψήφου. Ε, ίσως είναι κάποιο λάθος. Αν είναι δυνατόν πως μπορώ να, να πάρω και εγώ τον λόγο. Εγώ ζήτησα να πάρω τον λόγο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Για το προηγούμενο, για το προηγούμενο. Καλά μίληστε, καλά μίληστε. Και μετά θα ξεκινήσουμε για το επόμενο θέμα. Κύριε Τζαμπάφσκι, ε, σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω λοιπόν την επεξήγηση ψήφου μου για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή, γι' αυτό δεν μπορούσα να πάρω το λόγο Η μεταναστευτική κρίση στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι πρέπει να βρούμε μια συστημική λύση και εντός και εκτός της Ένωσης. Συνεργαζόμενοι με τις τρίτες χώρες ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παράτυπης μετανάστευση στις χώρες πρόέλευση δηλαδή. Να ε, δαπανίσουμε τους κατάλληλους πόρους για την ε, αντιμετώπιση ε, των, αιτίων αυτών. Το 5% το ανώτατο όριο δεν με ικανοποιεί. Εγώ γι' αυτό στην τελική ψηφοφορία δεν θα μπορέσω να στηρίξω την άποψη του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Και... Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση Φαγιών. Ο κύριο Τζαμπάσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα εγώ αυτή την έκθεση. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει ένα νέο ταμείο για την νέα πολυετή περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Πολύ ωραία όλα αυτά. Η δική μου χώρα, η Βουλγαρία, συνορεύει με μια χώρα που δεν θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τέρο μας, την Τουρκία δηλαδή. Ένα μόνο τώρα παράδειγμα θα σας δίνω των πρακτικών που ακολουθούνται και οι οποίες βαφτίζονται ως χρήσιμες, βοηθητικές πρακτικές. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην έκθεση αυτή είναι εντελώ αντιφατικοί ένας άνθρωπος ο οποίος παράνομα έχει μπει στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να έχει απαιτήσει όσον αφορά την άδεια παραμονής ή το άσυλο τη στιγμή που παράτυπα και παράνομα έχει μπει στη χώρα αυτή. Ο κύριος Σκούτσικ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε ότι η πολιτική μας για την προστασία των ε, εξωτερικών συνόρων γίνεται μέσω της ολοκληρωμένης προστασίας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με βάση τις σωστές δικλείδες ασφαλείας, παράλληλα με την ελεύθερη διακίνηση, κυκλοφορία των ατόμων εντός της Ένωσης. Ένα βασικό συστατικό της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση για να δημιουργηθεί αυτό το μέσο για την οικονομική στήριξη, για την διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις. Είμαι υπέρ του χρηματοδοτικού αυτού πλαισίου που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις εξελισσόμενες προκλήσεις πιο αποτελεσματικά. Είναι ένα σωστό βήμα προς την ουσιαστική διαχείριση και την ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πόλτσακ, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί ο χώρος έγκαιν και η ύπαρξή του είναι κάτι που θεωρώ είναι θεμελιώδες επίτευγμα της Ένωσης. Οπότε η έκθεση αυτή είναι ένα παραπάνω βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κοινή διαχείριση των συνόρων με επαρκή χρηματοδότηση είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως οι μεταναστευτικές ροές που εξακολουθεί να είναι θέμα. Οπότε λυπάμαι που το μέσο αυτό ε, δεν ενεκρίθη πλήρω, γιατί θα μας επέτρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τη συνεργασία των συνοριοφυλακών με τις αστυνομικέ αρχές, αλλά είναι καλό βήμα και γι' αυτό το υποστήριξα. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση Χολμάιερ. Η κυρία Μακοβέ έχει το λόγο. Μόνικα. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ταμείο εσωτερική Ασφάλειας. Ξεκίνησε το 2014 για να διευκολύνει την διασυνορική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το ταμείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του και θα χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια για την επόμενη οικονομική περίοδο 2021-2027 γιατί η εσωτερική ασφάλεια και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους τους ευρωπαίου πολίτες. Το οργανωμένο, διασυνορικό οργανωμένο έγκλημα έχει αυξηθεί τελευταία μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα κονδύλια είναι απαραίτητα για να ασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και προκειμένου να αγοραστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα βοηθήσει να σκανάρονται τα διαβατήρια όλων των ατόμων τα οποία διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σκανάρετε και το πρόσωπο των επιβατών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό το ταμείο θα χρειαστεί για τον καινούργιο εξοπλισμό. Δυστυχώς ε, δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη πρόσβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στη συντολογική σα ψήφου όσον αφορά τι προτάσει ψηφίσματο Μια ευρώ προστατεύει καθαρό αέρα για όλου. Ο κύριο Νέκοβ για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στήριξα, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί θεωρώ ότι το περιβάλλον εκείνη μα ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να δίδουμε το παράδειγμα. Δυστυχώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, η Σόφια, η πρωτεύουσα της δικής μου χώρας, βρίσκεται στην θέση υπαριθμών 15 σε ό,τι αφορά την μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλο τον κόσμο. Ε, βασική αιτία είναι τα συστήματα θέρμανσης. Επίσης έχουμε πολλά παλιά αυτοκίνητα, το σύστημα το μέσο μαζικής μεταφοράς είναι πεπαλαιωμένο επίσης, και προφανώς έχουμε και μόλυνση από τις βιομηχανικέ καταστάσει. Όλα αυτά θα πρέπει να καταπολεμηθούν ταυτόχρονα με την έλλειψη κατανόησης και τη φτώχεια. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να αποφύγουμε ε, περαιτέρω επενδύσεις στην υγεία. Η κυρία Κρούπα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ απήχα από την ψηφοφορία για το ψήφισμα αυτό. Μια ευρώ προστατεύει καθαρό αέρας για όλους. Σαφώς υπάρχουν σοβαρότα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, αλλά είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να αναβάλουμε οποιαδήποτε έμπρακτη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030 και να λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εντελώ από το 2030 και μετά να χρησιμοποιούμε άνθρακα. Στην Πολωνία, το μεγαλύτερο τμήμα τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια βασίζεται στον άνθρακα. Επομένω, δεν μπορούμε εμεί να ακολουθήσουμε τη δράση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και μέσω των ορεικτών καυσίμων να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συνδυάσουμε τώρα την προμήθεια σε ενέργεια, με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, βλέπουμε ότι τα δύο αυτά δεν παντρεύονται. Υπάρχουν πολλέ έρευνε οι οποίε προσπαθούν να προωθήσουν τι καινοτόμε μορφέ τη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και για επίπεδα πάνω από 20 ΜΒ την ώρα. Και προσπαθούν να μειώσουν επίση τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Κυρία Σπυράκη έχει το λόγο για ένα λεπτό ψήφισα τη στρατηγική για τον καθαρό αέρα παρά τις αντιρρήσεις του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος για δύο σοβαρούς λόγους. πρώτα απ' όλα τα εθνικά ανώτατα όρια για τους έξι βασικούς ρήπους που καταστρέφουν την υγεία μας την υγεία των πολιτών και προκαλούν πολλές ασθένειες μειώνονται. δεύτερον γιατί η ρήπανση όπως ξέρετε δεν ξέρει σύνορα δεν γνωρίζει σύνορα και γι' αυτό οφείλουμε να επιμείνουμε οι διεθνείς κανόνες για τη διακρατική ρήπανση να έχουν ακόμη μεγαλύτερη απέτηση από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης. κυρίως όμως πρέπει να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και τις τοπικές αρχές ώστε να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και να αντικαθιστούν παλιά οχήματα με τη συμβολή της ευρωπαϊκής ένωσης το παράδειγμα προς αποφυγή σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο του οαστ στη θεσσαλονίκη λεωφορεία που μολύνουν τον αέρα μας δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και αντί επενδύσεων σε νέα οχήματα μόνο προεκλογικές προσλήψεις. σας ευχαριστώ πολύ. Σαφώ θα πρέπει να αποτελέσει η πρωταρχική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα με τι απαιτήσει μα. Η ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε ότι τα πρότυπα δεν τηρούνται, ιδίω όσον αφορά τα σωματίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα εισάγοντα νέου κανονισμού, πολλού διαφορετικού κανονισμού νέους περιορισμούς όσον αφορά τη μόλυνση και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως εκταμιεύει και πάρα πολύ σημαντικά ποσά και δημιουργεί ταμεία, αλλά η ποιότητα του αέρα δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν δεν υπάρχουν κοινέ συντονισμένε προσπάθειε. Δεδομένου ότι υπάρχουν τρίτε χώρε αλλά και ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν δεόντω του κοινοτικού κανονισμού. Θα πρέπει να εξορροπήσουμε σωστά τη δράση και τις ε, κοινωνικές δαπάνες, τις κοινωνικές επιπτώσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε επίσης τον αέρα από την εθαλομίχλη προκαλείται από τα φτηνά μέσα θέρμανσης. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε ώρα πάνω από 700 άτομα χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ρήπανσης αυτής. Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι εκτεθειμένο στον, στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρόωρων θανάτων και χάνονται, χάνουν τη ζωή τους πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλά βρέφη. Καταλαβαίνετε ότι οι αριθμοί πολλές φορές είναι πιο ανησυχητικοί και πιο τρομακτικοί από την ίδια την ελονοσία ή από τους ίδιους τους πολέμους. Α μην ξεχνάμε τι είπε ο κύριο Τραμπ όταν αποχώρησε από τη Συμφωνία των, Παρουσί... των Παρισίων. Είπε ότι δεν μπορώ εγώ να ακολουθήσω τους στόχους του Πίτσμπρουκ. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικά αδιανόητο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταβάλουμε συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κυρίως για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο εκείνο που θα πούμε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι πιο σημαντικό και από την πυρηνική απειλή. Ο κύριο Λέρνερ έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Η κυρία Λέρνερ, συγγνώμη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Η καλή ποιότητα του αέρα είναι θεμελιώδε θέμα για όλου μας. Γι' αυτό ήταν πολύ σαφέ ότι θα υπερψήφιζε αυτή την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ψήφισμα αυτό ασχολείται με ε, ρηπαντές και την ποιότητα του αέρα και εντός των κτηρίων γιατί πολλοί ε, βεβαίως περνάνε πολύ καιρό εντο των κτηρίων όπου η ποιότητα του αέρα μπορεί να είναι χειρότερη από ότι στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αλλιώ πολλοί αρρωσταίνουν τόσο πολύ που την υπόλοιπη ζωή του ε, αντιμετωπίζουν ασθένειε που προκλήθηκαν από το χώρο εργασία του πολλοί υφίστανται και στα σπίτια τους και στους χώρους εργασίας ε, τις συνέπειες της κακής ποιότητας του αέρα. Πολλοί έχουν χάσει τη δυνατότητα να εργάζονται πλέον. Έχουμε πολλά προβλήματα και με την υγρασία που είναι πρόβλημα σε πολλούς χώρους εργασίας ή και σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής παιδιών και διαμερίσματα ο καθαρός αέρας. Είναι σημαντικό τμήμα της υγείας και ε, της ευημερίας όλων μας. Γι' αυτό είμαι υπέρ οποιασδήποτε δράση για να βελτιωθεί ποιότητα του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση Φώτιγκα. Γύρι Πάινεν, παρακαλώ, για ένα λεπτό. στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε, βλέπουμε φαινόμενα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να κάνουμε κάτι. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε πλέον ότι θα αναλάβει μια ε, κανονιστική προσέγγιση ε, και θα ε, επιβάλλει περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θεμελιώδες όμως πρόβλημα είναι να αποφασίσει κανείς τι είναι προπαγάνδα. Πώς θα την ορίσουμε και ποιος θα το κρίνει αυτό. η διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό είναι πολύ δύσκολη να γίνει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα μέσω του νόμου. Μία είναι η λύση. Ας μάθουμε από την αρχαία Ελλάδα δίκαιη και ισότιμη συζήτηση, ο ισότιμο διάλογο είναι ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την πρόταση, διότι ε, δεν είναι αντίθετη με το πνεύμα τη αλεύθερη και δίκαιη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Τώρα, όσον αφορά τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μονακό, τη Ανδόρα και του Αγίου Μαρίνου, έκθεση Λόπε Αγκουιλάρη. Κυρία Κέντζ έχει το λόγο. Παρακαλώ, Σεσίλ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την ψηφοφορία αυτή επιβεβαιώνεται κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία που μας δώσαν η, διαπραγματευ... η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με την Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και καταφέραμε να ενισχύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ολοκλήρωσής του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φίλοι μας από τον Άγιο Μαρίνο βρίσκονταν πάντα στο κέντρο της ευρωπαϊκής ιστορίας και η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται ανέκαθεν στις κοινέ πολιτιστικές αξίες που έχουμε έχουμε με τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον πριν το τέλος της θητείας αυτής, να έχουμε μια κοινή πολιτική δήλωση, όπου θα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές το συντομότερο δυνατό και δυνατόν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Διακόπτεται τώρα η συνεδρίαση και θα συνεχιστεί στις 3 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.